θέμα την ε, προφορική απάντηση στο ερώτημα για την ε, διαχείριση του τομέα της ζάχαρης ε, σήμερα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους συντάκτες της ερώτησης. Ε, πρώτη ομιλήτρια θα είναι η κυρία Γιανακουδάκη. Κυρία Επίτροπε, κάθε φορά που ζητούμε από σας να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό, από σας, από την Κομισιόν, παίρνουμε την ίδια απάντηση. Μας λέτε δεν υπάρχει πρόβλημα. Κι όμως οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας Ζάχαρο Κάλαμου αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες. Τα εργοστάσια κλείνουν για αρκετές μέρες την εβδομάδα και αυτό σημαίνει ότι χάνονται και θέσεις εργασίας. Η Κομισιόν μας έδειξε μάλιστα αντίγραφο παραγωγό από τη Γαλλία που έλεγε ότι ανέκαθεν οι προμήθειες δεν έφθαναν και ότι παρόλα αυτά επιμένεται να διατηρείται την κατάσταση ως έχει. Αυτό το οποίο σας ε, διέφυγε είναι ότι η εγκατάσταση αυτή ανήκει σε πραγωτεύθλων. Πότε θα παραδεχθεί η Επιτροπή ότι υπάρχει πρόβλημα ή θα μας πει ότι είναι μόνο βρετανικό πρόβλημα. 62 βουλευτές από 11 χώρες έγραψαν στον Επιτροπό Υπεύθυνο για τα θέματα Γεωργίας και ζήτησαν αλλαγές στο καθεστώς της ζάχαρης κινδυνεύουν θέσει εργασία, όχι μόνο στον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, τη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Το γνωρίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα, κύριε Επίτροπε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα οι κανόνε να ισχύσουν για όλου με τον ίδιο τρόπο. Κύριε Επίτροπε, δεν είστε υπεύθυνοι για τα θέματα γεωργία, αλλά για τα θέματα των Ευρωπαίων πολιτών, του οποίου καλείστε να υπερασπιστείτε. Υπάρχουν λοιπόν θέσει εργασία που απειλούνται όπω είπα και επιπλέον όλοι σε λίγο θα πληρώνουμε την ζάχαρη πιο ακριβά τη στιγμή που ήδη είναι ακριβότερη κατά 46% σε σχέση με την παγκόσμια αγορά. Α δούμε λοιπόν την πηγή του προβλήματο. Α δούμε το πρόβλημα του εφοδιασμού και στο λύσουμε. Αν μα πείτε και πάλι όχι, θα απαγοητεύσετε του ανθρώπου του οποίου υποτίθεται ότι υπηρετείτε. Και οι Ευρωπαίοι, η Ευρώπη εν γέννη θα χάσει άλλη μία με ποιητική βιομηχανία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λάν είναι επίση συντάκτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω, θα ελπίζω ότι η Επιτροπή Γεωργίας θα ήταν εδώ για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Αλλά ξέρω ότι κάνετε μια πολύ καλή δουλειά και θα προσπαθήσετε να απαντήσετε. Η συζήτηση εστιάζεται στην ε, διαχείριση του ε, της ε, ζάχαρης. Ε, η πρόβλεψη της Επιτροπής του 2006 για τις εισαγωγές από τις χώρες ΑΚΕ τελικά δεν εκπληρώθηκε και η Επιτροπή αρνήθηκε να κάνει εισαγωγές από άλλες χώρες όπως είναι η Βραζιλία για να δισταθμίσει αυτή τη διαφορά. Με τον τρόπο αυτό εκτινάχθηκε το κόστος για τις πρώτες ύλες ε, μειώθηκε η παραγωγή, αυξήθηκε το κόστος και τελικά ε, οι τιμές ε, της ζάχαρης από ζαχαράτευτολα δεν είναι πλέον ανταγωνιστικές, ε, από δεν είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με τη ζάχαρη από ζαχαρά Ε, με τον τρόπο αυτό απολέστηκαν, θα απολεστούν πάρα πολλέ θέσει εργασία σε πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θέλουμε είναι θεμητό ανταγωνισμό, ισότιμοι όροι και η Επιτροπή εμποδίζει να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν επιχειρήματα από τις παραγούς ε, Ζαχαρότευτλα ε, που, ανα... λένε ότι έχει εκπληρωθεί η εξαγγελία της ε, Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να προσέξει στις εισαγωγές από την Βραζιλία. Επίσης λέει ότι είναι αποτυχία του τομέα του ζαχαρακάλαμου που δεν μπόρεσε να προβεί σε αναδιάρθρωση και αυτή είναι η ουσιαστική αιτία του προβλήματος. Έτσι λοιπόν το ζήτημα είναι ποιο έχει δίκιο και τι δράση θα πρέπει να αναλυφθεί. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία κατά την άποψή μου ότι υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα στο τομέα του ζαχαρακάλαμου. Και θα ήθελα να ακούσω από τον Πίτροπο σήμερα τι δράση θα αναλάβει για να εξασφαλίσει ισοτιμία των όρων ε, μεταξύ παραγωγών ε, ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είναι η κυρία... θα πρέπει να ρωτήσω την κυρία Γιανακουδάκη εάν ε, θέλει να απαντήσει σε δύο ερωτήματα των συναδέλφων τα οποία μόλις έλαβα αλλά τα οποία απευθύνονται στην κυρία Γιανακουδάκη. Ε, συμφωνείτε κυρία Γιανακουδάκη με αυτά τα δύο ερωτήματα. Εάν ε, συμφωνείτε θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Μωράης να υποβάλει το πρώτο ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και κυρία Γιανακουδάκη. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Εγώ στο Λονδίνο έχω ένα σημαντικό εργοστάσιο ζάχαρης. Διάφορα μέτρα λήφθησαν τα τελευταία δύο χρόνια για να εξασφαλίσουν τον ομαλό εφοδιασμό των εργοστασίων και αυτό ως τώρα έγινε με τους ίδιους όρους για όλων των μορφών πρώτη ύλη. κουδάκι, οι δεσμοί για την ισογλυκόζη και τα τέφτλα ήταν 75 ευρώ ανατόνο για 1,2 εκατομμύρια τόνους. Για την ακατέργαστη ζάχαρη, λιγότερα από 900.000 τόνοι εισήχθησαν και ο μέσος δασμός ήταν γύρω τα 183 ευρώ ανά τόνο. Αυτά είναι τα νούμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Το δεύτερο ερώτημα είναι από τον κύριο Ταραμπέλα προς την κυρία Γιάννα Κουδάκη. Κυρία Γιάννα Κουδάκη, αυτή συναδελφή, εξεπλάγει από την αδικαιολόγητη επίθεση σας κατά της Κομισιόν, γιατί αν κατάλαβα καλά μας λέτε για δυσκολίες, θα συγκινηθούμε για τις θέσεις που θα χαθούν, όμως το 2006 δεν θυμάμαι να επαναστατήσετε, γιατί η μεταρρύθμιση του 2006 άλλαξε τον τομέα, κάποιοι δεν άλλαξαν, βιομηχανίε που αρνήθηκαν να αλλάξουν και των οποίων υπεραμείνεστε. Και θέλω πραγματικά να σα ρωτήσω αν εφαρμόζετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, δεν καλέσετε κάποιου να αναδιαρθωθούν και ξαφνικά τώρα τα λόμπι σα πιέζουν να μα πιέσετε. Κύριε Γιανακουδάκη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε κανένα. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θέλουμε ένα ισότιμο πεδίο. Μιλούμε για ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας. Τώρα το 2.006 θα ε, και μια νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνη την εποχή ήταν λογική και κατά πάσα πιθανότητα δούλεψε. Αλλά οι επιχειρήσεις ε, και τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξελιχθούν καθώς οι καταστάσει αλλάζουν και οι καταστάσει πράγματι άλλαξαν και η ζάχαρη πλέον δεν επαρκεί για τις ε, μονάδες ε, κατεργασίας και έπρεπε να κλείσουν ορισμένε μέρε τη εβδομάδα. Αυτό είναι γεγονός. 4.500 ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας θα απολεστούν και μιλώ για θέσεις εργασίας όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε χώρες όπως είναι η Πορτογαλία που πραγματικά υποφέρει τρομερά από την ύφεση. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να παίζουμε με την πολιτική. Ε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή ακούμε τις, ε, τους συντάκτες δεν έχουμε προχωρήσει πραγματικά στη συζήτηση και θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι συντάκτες του ερωτήματος ε, παρουσιάζουν το ερώτημα που έθεσαν προς την Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά έχω και μία άλλη μπλε κάρτα ε, η οποία απευθύνεται επίση προς την κυρία Γιάννα Κουδάκη. Είναι της, εκ της κυρίας Πατράου. Ε, θα, τη δεχτείτε? Ναι, παρακαλώ. De Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο μιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, δεν είχε ανοίξει το μικρόφωνο μου. Μετά από όσα 20 άκουσα, αισθάνομαι την υποχρέωση να ρωτήσω το εξή. Εμεί έχουμε μια βιομηχανία που δεν έχει πρώτε ύλε για να εργαστεί. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβλέψει εισαγωγέ ε, με αξία 6,3 ε, εκατομμυρίων τόνων και ε, τώρα προβλέπονται μόνο ένα εκατομμύριο τόνοι για τις εισαγωγές ε, και θα ήθελα να ρωτήσω μια τόσο μικρή ποσότητα η οποία δεν επαρκεί για τη βιομηχανία μας ή διασφαλίζεται διότι δυστυχώς πρέπει να το θέσουμε και αυτό εδώ στην Ολομέλη. Ευχαριστώ. Κυρία συνάδελφε. Συμφωνώ πολύ τους μαζί σας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας και αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε τώρα. Γι' αυτό προσπαθούμε να δράσουμε. Οι δυνατότητες ε, σημαντικής ε, αύξησης της ποσότητας από προτιμησιακή προμήθειες είναι πολύ μικρή, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει μια απάντηση στη συγκεκριμένη κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, συνεχίζουμε με τις ε, ομιλίες, με τις παρεμβάσεις των συντακτών του ερωτήματος. Ο κύριος Καπούλα Σάντος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω διότι ο Επίτροπος Γεωργίας φάνηκε διατεθειμένος να συζητήσει για τις ε, διάφορες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα. Κυρία Επίτροπε όμως, δεν φτάνει μόνο να γίνει ο διάλογος ε, εάν δεν υπάρχουν αποτελέσματα ε, και αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Είναι αλήθεια κύριε Επίτροπε ότι μετά από τη μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης το 2006 τα εργαστήρια επεξεργασίας ζάχαρης ε, ε, δια, έχουν όλο και σοβαρότερα προβλήματα για την εξέβρεση πρώτη ύλη την οποία θα πρέπει να κατεργαστούν. Ε, τα όσα αποφασίστηκαν το 2005 ε, βασίστηκαν σε λανθασμένες εκτιμήσεις και στη συνέχεια έγιναν και άλλες εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες. Μπορώ να δεχτώ όλα τα επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης της ευρωπαϊκής παραγωγής, διότι αυτό μας ενδιαφέρει. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως μεταξύ των οποίων και στην Πορτογαλία, έχουμε οικονομίες οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό ε, στην ε, δυνατότητα να έχουμε εισαγωγή ε, ζάχαρης από ζαχαροκάλαμα και δεν μπορούμε να πούμε στον κλάδο ότι το πρόβλημα πρέπει να το λύσουν μόνοι τους. Ε, γνωρίζουμε όλοι ότι οι οικονομικοί παράγοντες λαμβάνουν αποφάσεις βάσει των όσων προβλέπει ο Ευρωπαίος Ρυθμιστής. Και αυτό που ισχύει όμως και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σε αυτή την περίπτωση δεν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις που θα επιτρέψουν να υπάρχει ισορροπημένη συνεργασία μεταξύ των τομέων που έχουν πρόσβαση στην αγορά και να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ε, τη συνέχεια των 250.000 ε, ε, θέσεων εργασία στον τομέα τη ζάχαρη στην Ευρώπη, κάτι το οποίο είναι κεφαλαιόδη σημασία στου χαλεπού κυρίου. Τώρα θα έρθουμε στον τελευταίο συντάκτη του ερωτήματο, τον κύριο Αλφρετ Ρούμπιξ. Πρόεδρε, Η ουσία του προβλήματος είναι η εξή. Η μεταρρύθμιση είχε αποτέλεσμα να γίνουμε καθαρή εισαγωγή από εξαγωγή. Πολλοί παραγωγοί πιστεύουν ότι φταίει το σύστημα ποσοστώσεων, το οποίο οδήγησε στην καταστροφή πολλών βιομηχανιών ζάχαρης. Στην Λετωνία τρία εργοστάσια έκλεισαν λόγω των ποσοστώσεων. Οι παραγωγοί ζητούν επανεισαγωγή του παλιού συστήματος. Το ίδιο συνέβη και στη Γερμανία. Οι Γερμανοί παραγωγοί μου έστειλαν επιστολή με την οποία ζητούν την επαναθέσπιση του παλαιού καθεστώτος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να καταργηθούν οι ποσοστώσει. Χάσαμε το 80% του παραγωγικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σας πω. Το σύστημα λοιπόν πρέπει να παραμείνει ως έχει ω το 2020. Το σημερινό σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Γνωρίζουμε το κόστος της παραγωγής ένα εκτάριο. Ξέρουμε λοιπόν που πηγαίνουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να στριμώξουμε περαιτέρω τους παραγωγούς. Ας κοιτάξουμε να κάνουμε κάτι για τις τιμές. Για να μπορέσουμε να είμαστε και ανταγωνιστικοί στην αγορά. Η σημερινή πολιτική δεν θα επιτρέψει στον τομέα της ζάχαρης να αναπτυχθεί. Ας υποστηρίξουμε λοιπόν καταρχήν την παραγωγή και τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα περάσουμε τώρα στην απάντηση εκ μέρους της Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του συναδελφού Τσόλεος, θα προσπαθήσω να απαντήσω στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι η μεταρρύθμιση του Νοεμβρίου του 2006 της κοινή οργάνωσης αγοράς της ζάχαρης είχε ως στόχο να κάνει τον τομέα πιο ανταγωνιστικό. Ο τομέας του τεύτλου λόγω του κλεισμένου πολλών εργοστασίων ούτως ή άλλως αντιμετώπιζε προβλήματα και στον τομέα του ζαχαροκάλαμου την εποχή εκείνη χρειαζόταν 150 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει ανταγωνιστικός. Την εποχή εκείνη απαλείψαμε τη διαφορά μεταξύ των παλαιών των παραδοσιακών και των νέων παραγωγών με μεταβατική περίοδο τριών ετών που εξέπνευσαν το 2009. Παραλλήλως, η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίσε πρόσβαση χωρίς δασμούς στις χώρες ΑΚΕ με ρήτρα διασφάλισης όμως στην περίπτωση που οι εισαγωγές θα ξεπερνούσαν τα 3,5 εκατομμύρια τόνους. 1,6 από τις χώρες ΑΚΕ. Στην συνέχεια μειώσαμε τις εξαγωγές σε 1,35 εκατομμύρια τόνους. Μετά από την μεταρρύθμιση η ποσόστοση μειώθηκε σε 13,5 εκατομμύρια τόνους σε σύγκριση με τα 17,4 εκατομμύρια τόνους το 2004-2005. 41% λοιπόν των εργαστοσίων έκλεισε. Εκ παραλλήλου, το δυναμικό επεξεργασίας από 1,5 εκατομμύρια τόνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε στα 27. Και η παραδοσιακή παραγωγή από 1,15 εκατομμύρια τόνους ανέβηκαν κατά πολύ. Οι σημερινές εισαγωγές γίνονται με βάση προτιμησιακές συμφωνίες με τις χώρες ΑΚΕ και με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 1,8 εκατομμύρια συγκεκριμένα τόνοι φέτος. Σύνολο λοιπόν μαζί με, τη, με τις 670.000 τόνους και τους 380.000 τόνους από τα Βαλκάνια και τους 400.000 τόνους από τους ε, διαγωνισμούς. Φτάνουμε στα 3,2 συνολικά εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Για του χρόνου 300.000 τόνοι θα δοθούν στην Νότιο Αμερική και επιπλέον 400.000 τόνοι ζάχαρης εισάγονται κάθε χρόνο, κάθε χρόνο με την μορφή μεταποιημένων προϊόντων. Η περίοδος 9-10 δεν ήταν σαν τις άλλες. Η τιμές στην παγκόσμια αγορά ήταν υψηλότερες από τις τιμές στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο ήταν χωρίς προηγούμενο τα τελευταία 50 χρόνια. Ως εξ αυτού οι χώρες ΑΚΕ προτιμήσαν να πωλήσουν στην παγκόσμια αγορά την παραγωγή τους ή στην εσωτερική αγορά και δεν έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προβλεπόμενα. Η ισορροπία λοιπόν στην ευρωπαϊκή αγορά κινδύνευσε αν και η μεταρρύθμιση ήταν σαφή. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση έχει την Κομισιόν η δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα για να εξορροπήσει λοιπόν την αγορά. Προ το σκοπό αυτό, η Κομισιόν κατά τη διάρκεια των περίοδων 10-11 και 11-12 εξασφάλισε, επέτρεψε μάλλον προτιμησιακέ εισαγωγέ για την εισαγωγή ποσοτήτων εκτός ποσοστώσεων με τρόπο συντονισμένο όσον αφορά τη συνολική ποσότητα αλλά και τους όρους. 2,35 εκατομμύρια τόνοι συνολικά εισήχθησαν επιπλέον και διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά. 1,25 εκατομμύρια τόνοι ήταν εισαγωγές. ορισμένη ορισμένη εργοστάσια παραπονούνται όντω για να υπάρχει εφοδιασμό και ορισμένοι από εσά έθεσαν ακριβώ το ίδιο ερώτημα. Τι σημαίνει όμω την πραγματικότητα. Πρώτη διαπίστωση. Η θέση αυτή δεν είναι θέση όλων των εργοστασίων ζάχαρη στην Ευρώπη. Δεύτερο γεγονό. Τι λένε τα νούμερα όσον αφορά τι εισαγωγέ. Πριν από την μεταρρύθμιση του 2005 εισάγαμε 2,3 εκατομμύρια τόνους. Μετά από την μεταρρύθμιση οι εισαγωγέ αυξήθηκαν. Τώρα λέει κανεί λοιπόν ότι εισάγουμε λιγότερη ζάχαρη, λιγότερη μάλλον ύλη και ότι κάποιοι έχουν δυσκολίε δεν είναι απλούστατα αλήθεια. Ποιο είναι λοιπόν το πραγματικό πρόβλημα. Μια δελεχιαστερή ανάλυση κατά κράτο μέλο και κατά εργοστάσιο καταδεικνύει ότι ο τομέας της επεξεργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, Άλλωστε αυτό επεδίωξε η μεταρρυθμίση του 2005, τον πραγματικό ανταγωνισμό. Ορισμένα κρατημέλη και ορισμένα εργοστάσια ζάχαρης αύξησαν το δυναμικό τους, τη δυναμικότητά τους, εξασφαλίζοντας προμήθεια πρώτης από τις τρίτες χώρες. Άλλα εργοστάσια συρρυκνώθηκαν παρά το γεγονό ότι η συνολική προμήθεια πρώτη ύλη για την Ευρώπη αυξάνεται. Πρόκειται λοιπόν για θέμα εμπορική στρατηγική ιδιωτικών επιχειρήσεων. Κυρίε και κύριοι, η επεξεργασία ζάχαρη στην Ευρώπη γίνεται πλέον με όρου παγκοσμίου εμπορίου μετά τη μεταρρύθμιση του 2005. Μετά από μια μεταβατική βεβαίω περίοδο, η οποία εξέπνευσε το 2009. Αυτό άλλωστε ήταν και η επιδίωξή μας. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Η Κομισιόν φροντίζει για την ισορροπία στην ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης. Οι εισαγωγέ αυξήθηκαν το από το 2006 και φτάσαμε στο ιστορικό υψηλό των 4 εκατομμυρίων τόνων το 2011. Οι εισαγωγές από τις χώρες ΑΚΕ ακολούθησαν την ίδια ακριβώ τάση. Αν οι χώρες ΑΚΕ αποφασίσουν να εξαγάγουν ραφιναρισμένη ζάχαρη ως τελικό προϊόν, αυτό δεν μπορεί να μας βρει αντίθετους. Το πρόβλημα λοιπόν δεν έχει σχέση με την έλλειψη ζάχαρης, αλλά με τον ανταγωνισμό μεταξύ ευρωπαϊκών βιομηχανιών, λόγω του κάποιοι μεταξύ άλλων αυξήσαν και την δυναμικότητά τους την δυναμικότητα επεξεργασία. Γι' αυτό και ορισμένα εργοστάσια δεν δουλεύουν στο 100% τη δυναμικότητά του. Ο βασικό στόχο τη μεταρρύθμιση του τομέα ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και ο επαναπροσανατολισμό τη Ευρωπαϊκή Βιομηχανίας Ζάχαρης προ την παγκόσμια αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθαρό αγωγέα πλέον, ενώ στο παρελθόν ήταν σημαντικό εξαγωγέα. Η μεταρρύθμιση λοιπόν αποτέλεσε επιτυχία διότι ακριβώς κατέληξε στο να μειωθεί η παραγωγή πλεονασματικής ζάχαρης. Αυτήν την στιγμή οι ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι το 2015. Τον Οκτώβριο του 2011 μάλιστα η Κομισιόν υπέβαλε πρόταση για την μελλοντική λειτουργία του τομέα της ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την οποία θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις παραγωγής. Αυτό είναι ακριβώς που συζητούμε αυτή τη στιγμή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εκ μέρους του συναδέλφου μου, του Επιτρόπου Τσιόλος, σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά στον διάλογο αυτό για την αγορά της ζάχαρης μέχρι το 2013 και την κατάργηση των ποσοστώσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό θα το κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει και το ερώτημα αυτό. Ε, και θα ήθελα ξεκινήσουμε τώρα την ε, συζήτηση με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Ντές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο σωλής εφοδιασμό τη Ευρωπαϊκή Αγορά με ζάχαρη θα πρέπει να είναι πρώτος στο στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής ζάχαρης. Με την ε, μεταρρύθμιση του κανονισμού το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο έγινε, άρχισε να εξαρτάται από τις εισαγωγές. Η κυρία Ρέντινγκ ε, ανέφερε αριθμούς. Ε, έγιναν απαραίτητες εισαγωγές αλλά λόγω κακής ε, εγκομιδής σε πολλές, σημαντικές, σε πολλές χώρες παραγούς της ζάχαρης τιμές έμειναν ε, πίσω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε κυρία Ρέντινγκ, έλαβε τα σωστά μέτρα. Διευκόλυνε τις εισαγωγές χωρίς δασμούς, πάνω 500.000 τόνους και έδωσε δυνατότητα στους εγχώριους παραγωγούς γλυκόζης και τέφτλων να μπορέσουν να πουλήσουν ένα τμήμα της παραγωγής τους στον, στην ευρωπαϊκή αγορά. Και σε αυτό το υπόβαθρο, με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η κυρία Ρέντινγκ ε, θα πρέπει να τύχει τη δική μας υποστήριξη. Ο κανονισμός για τη ζάχαρη διαθέτει τα αναγκαία εργαλεία για να εξασφαλίσει τον αφοδιασμό με ζάχαρη και να εξορπίσει σωστά τα διάφορα συμφέροντα. Και αν μιλούμε για την ε, απώλεια θέσεων εργασία στην οποία αναφέρθηκε η πρώτη αμιλήτρια, θα ήθελα να αναφερθώ στο όσα είπε και ο κύριος ε, Ταραμπέλα στην, ε, κατά τη μεταρρύθμιση της ε, αγοράς χάθηκαν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα στο Άνω Παλατινάτο ε, έκλεισαν πολύ σημαντικά εργοστάσια με χιλιάδες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό δεν είναι το να προβάλλουμε αυτό το επιχείρημα. Το ζητούμενο δεν είναι εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά η εξασφάλιση μιας ισορροπίας στην κοινή οργάνωση της αγοράς. Γι' αυτό είμαι υπέρ μιας παράτασης του σχεδιασμού καθεστώτος. Έχω μία μπλε κάρτα από την ε, ε, κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ντες, γιατί αν τις ψηλές τιμές ζάχαρης, δέχεται οι τιμές της ζάχαρης να είναι σε 6 cents πιο υψηλές από τις ε, τιμές ε, παγκοσμίω. Και αυτά δείχνει στην κρίση της ζάχαρης το 2010 δηλαδή οι τιμέ τη ζάχαρη στην Ευρώπη εκτενώσαν στα ύψη, ενώ οι τιμέ παγκοσμίω ε, μειώνονται. Ε, και πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά ε, εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης από ζαχαρότευτλα ε, κλείνουν ενώ στηρίζεται η παραγωγή από ζαχαρκολά ενώ στηρίζεται η παραγωγή της ζάχαρης από τα ζαχαρότευτλα. με την μεταρρύθμιση του 2006 και ήδη πριν οι τιμές των σαχαρότεφλων στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 40%. Δηλαδή οι παραγωγές σαχαρότεφλων ε, είχαν σημαντικές ε, απώλειες και είχαμε τεράστιες διακυμάνσεις των τιμών στη συνέχεια. Ε, και οι τιμές ήταν πολύ πιο υψηλές παγκοσμίως από ό,τι στην Γερμανία. Αυτό ήταν τότε το πρόβλημα. Ε, κυρία συνάδελφε, θα, θα ήθελα να σας πω ότι αν ε, στην Ευρώπη καταργήσουμε την, ε, την κοινή οργάνωση αγοράς της ζάχαρη, θα είμαστε πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις των τιμών της ζάχαρης στην Ευρώπη και η παραγωγή της ζάχαρης θα πληρώσουν ένα πολύ υψηλό τίμημα. Κύριε Σταραμπέλα, ευχαριστώ πολύ ε, πιστεύω ότι το ερώτημα αυτό υπαγορεύεται από, από τα μεγάλα συμφέροντα των παραγωγών. Η κυρία Ρέντινγκ εξήγησε πολύ καλά την θέση της Επιτροπής, δηλαδή να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό με ζάχαρη για τον καταναλωτή και προσπάθησε να διτηρήσει αυτή την ισορροπία στην αγορά ε, αντιδρώντας ε, με ταχύτητα. Εγώ είμαι υπέρ μιας έγκρισης των ε, ποσοστώσεων ε, γιατί βεβαίω έχουμε όλοι ανησυχίε ε, για τι απώλειε των θέσεων εργασία. Θα πρέπει να τι προσαρμόσουμε τι ποσοστώσει προ τα πάνω, ούτω ώστε να ελέγξουμε συλλογικά την παραγωγή ζάχαρη. Γιατί ε, εάν δεν υπάρχει τέτοιο έλεγχο, υπάρχουν παρεκκλήσει, υπάρχει, υπάρχει ανεξέλεγκτη του κόστου που ζημιώνουν τους παραγωγού. Ε, νομίζω ο παγκόσμιος έλεγχος είναι ε, θεμελιώδης και θεωρώ ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε αυτές τις ποσοστώσεις για να αναζωογονήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία, τους ευρωπαίους ε, παραγωγούς. Ευχαριστούμε πολύ η κυρία Πρίτα Ράιμας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να πω ότι με τελευταία μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης πραγματικά χαράξαμε ένα σωστό δρόμο. Η βιομηχανία προσαρμόστηκε αντίστοιχα στην αγορά, αλλά τα παράπονα από πλευρές δείχνουν ότι θα πρέπει να εξελιχθούμε περαιτέρω, να εξελίξουμε περαιτέρω την αγορά ζάχαρης, γιατί οι προγνώσεις ε, κομισιόν δεν εκπληρώθηκαν, οι χώρες ΑΚΕ δεν ε, εξήγαν τη δική του ζάχαρη στην Ευρώπη, αλλά σε άλλες περιοχές του κόσμου, γιατί υπήρξε μια αλλαγή παγκοσμίως όλων των αγορών και εντελώς διαφορετικά από ό,τι είχε προβλέψει κανείς. Η ζήτηση ε, αυξήθηκε σε πολλές χώρες κατά το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει το παρελθόν. Η ζήτηση σε ζάχαρη αυξήθηκε παγκοσμίω και ε, ε, συνεπία αυτών των ε, τάσεων συρρυκνώθηκε η ευρωπαϊκή αγορά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε μόνο τη ζάχαρη ως προϊόν, αλλά ήδη η παραγωγή προσαρμόζεται στην αγορά και κάνουν, προχωρούν σε εναλλακτικέ μορφές παραγωγής. Για παράδειγμα, στη Γερμανία η παραγωγή ενέργειας ε, γίνεται στα χωράφια, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και αυτό, αυτός ο προγραμματικός ανταγωνιστής προς την ε, καλλιέργεια ζάχαρης από ζαχαρότευτλα. Ε, εγώ είμαι υπέρ της ε, άρσης των, του καθεστώτος των ποσοστώσεων. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριο Τζέιμς Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καλή η συζήτηση σήμερα το απόγευμα, παρά το γεγονός ότι είμαστε λίγοι. Ε, είναι και πολύ επίκαιρη η συζήτηση και συγχαίρω τους συναδέλφους που επέστησαν την προσοχή μας στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης του καθεστώτος της ζάχαρης ε, το 2006 αποδείχθηκε λανθασμένη. Αυτή τη στιγμή τα εργαστάσια κατεργασίας ε, ζάχαρης ε, βρίσκονται στην ανάγκη να εισάγουν ζάχαρη όπως ακούστηκε σήμερα και δεν νομίζω ότι ε, είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να ασχοληθούμε επίσης και το θέμα της ποιότητας μεταξύ των διαφόρων τύπων παραγωγής ζάχαρης. Για παράδειγμα, τα εργοστάσια κατεργασίας ζαχαροκάλαμου αντιμετωπίζουν προβλήματα για την προμήθεια πρώτης ύλη παρά τα όσα λέμε εμείς. θα δώσει λοιπόν στον κλάδο Ελλάδο τη λύση για τους δασμούς που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, διότι πραγματικά χάνονται θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους πολιτικής ομάδας είναι ο κύριος Αγνίου Τζον Στιούαρτ πρέπει να συγκρίνουμε τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους ευρύτερους στόχους πολιτικής για την απασχόληση, τις ε, κοινωνικές συνθήκες εργασίας και το εμπόριο και το τι λένε για τη ζάχαρη. Προσφάτως και ο Πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόζο και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Φανορόμπαη, μίλησαν σε ένα συνέδριο και ε, για την απασχόληση και επισήμαναν πόσο σημαντική είναι η ανεργία για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για τη ζάχαρη δεν ανέφεραν ότι η Ισλανδία, ε, η Νορβηγία και η Ελβετία έχει μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Ε, δεν κάνουν τίποτα για την ε, απασχόληση στην πραγματικότητα παρά το γεγονός ότι τη συζητούν συνέχεια. Υπάρχουν περιορισμοί στην προμήθεια ζάχαρης και αυτό είναι άμεση συνέπεια απώλειας θέσεων εργασίας στον τομέα της ζάχαρης. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι δασμοί βασίζονται σε ανακριβείς υπολογισμούς που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005 για τη ζάχαρη. Αν πραγματικά η ζάχαρη πρέπει να είναι λοιπόν σε προσεκή τιμή και θέλουμε να έχουμε θέσεις εργασίας, γιατί γίνεται αυστηρότερη, ακριβότερη συγγνώμη, προμήθεια ζάχαρης. Ο Επίτροπος Ντεγκούχτ προσφάτω αναφέρθηκε στην ανάγκη να αυξήσουμε το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε το ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με ε, ε, επί τον προϋπολογισμό μιας χώρας ε, όπως της Αδανίας ή της Αυστρίας η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν ρωτήθηκε για το τι θα κάνει ήταν να αναφερθεί στις διμερείς διαπραγματεύσεις που κάνουμε χώρες της κεντρικής αναφοράς. Ε, ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε ε, συμφωνίες ε, για τη ζάχαρη που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουμε από τις χώρες ακές και τις πιο ευγάλωτες ε, χώρες. Όσο πιο σύντομα λοιπόν αντιμετωπίσει το γεγονό ότι έχουμε απώλειες αυτή τη στιγμή στο θέμα τη ζάχαρη, ε, τόσο ε, καλύτερο θα είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το καθεστώ τη ζάχαρη. Κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ερώτηση ε, και θα έπρεπε αυτό να μα αφυπνήσει και να ξυπνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αντιληφθεί επιτέλου ότι υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω στον κύριο Νίκολσον γιατί όταν κάλεσα τον κύριο Άγνιου να πάρει το λόγο είδα ότι ε, σας απευθύνθηκε μία μπλε κάρτα. Την δέχεστε κύριε Νίκολσον από την κυρία Γιανακουδάκη. Ευχαριστώ. Δεν είναι φιλική αυτή η μπλε κάρτα. Δυστυχώς Έχω πάρα πολλέ ε, ερωτήσει που δεν απαντήθηκαν. Δεν φταίει η κυρία Ρέντινγκ βέβαια που χρειάστηκε να διαβάσει ε, μία ομιλία, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στου συναδέλφου ε, που ασχολούνται με θέματα γεωργία. Πριν από μερικέ εβδομάδε συναντηθήκαμε με τον Επίτροπο Τσόλο και του ζητήσαμε να καθορίσει μία task force. Έχετε κάποια νέα, θα αποκολουθήσουμε αυτή την άγουσα, ο κύριο Νίκολσον. Χαίρομαι που μιλώ αμέσως μετά από τον κύριο Άγνιου, ο οποίος σήμερα ε, ε, διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν ε, πρόφερα σωστά το όνομά του. Νομίζω ότι το είπα σωστά αυτή τη φορά. Να σας πω κυρία Γενακουδάκη ότι δεν έχω μάθει κανένα νεότερο, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή άγουσα. Δεν μπορούμε να πιστοχωρούμε, πρέπει να κοιτάμε προς το μέλλον, πρέπει να λησμονήσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος και να κοιτάξουμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Τσάου Φερέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, η τελευταία μεταρρύθμιση της αγοράς ε, ζάχαρης ε, κατέστρεψε την ε, βιομηχανία επεξεργασίας ζαχαρότητα στην Πορτογαλία και ένα μεγάλο τμήμα της ζήτησης μέχρι τώρα καλύπτεται από την εχόρια παραγωγή. Σήμερα είμαστε εξαρτημένοι από τις ε, ε, παγκόσμιες, ε, από την εξέλιξη παγκοσμίω των τιμών. Ε, πολλές, ε, πολλά εργοστάσια δεν μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν γιατί δεν έχουν τις πρώτες ύλες. Η Επιτροπή είναι συνυπεύθυνη για αυτές τις εξελίξεις και δεν είναι δυνατόν να συγκαλύπτει ή να αγνοεί αυτά τα προβλήματα γιατί οι προβλέψεις Επιτροπής δεν ανταποκρίθηκαν στην ζήτηση των εργοστασίων. Ε, θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι ποσοστώσεις ούτως ώστε να μπορεί κάθε χώρα να αξιοποιεί το εφιστάμενο δυναμικό της για την παραγωγή της ζάχαρης. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ελλείμματα σε εισαγωγή από ζαχαροκάλαμο και τα εργοστάσια δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να λειτουργούν дълго изказване, което вие ни прочетохте и му кажете да спре да играе игрички с нас, защото... Να πείτε στον Επίτροπο Τσιόλος, ο οποίο έγραψε τον λόγο σα, να σταματήσει να παίζει. Διότι αυτά τα παιχνίδια έχουν ω αποτέλεσμα να κινδυνεύουν εκατοντάδες χιλιάδε θέσει εργασία. Κάποιοι θα πεινάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι αρκούν δηλώσεις περί βελτίωσης της κατάστασης και ότι πλησιάζουμε στην παγκόσμια αγορά κλπ. Όταν ο μισός τομέας απολαύει προστασία και ο άλλος μισός έχει διαλυθεί. Η σημερινή συζήτηση κοντεύει 11 ίσα ίσα πρέπει να δείχνει ακριβώς πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε απάντηση. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το θέμα επιτέλους στα σοβαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μια μπλε κάρτα για σας. Την δέχεστε. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Πρόεδρε, ο κ. Στογιάννοφ θα μπορούσε να μας εξηγήσει ποιες θέσεις χάθηκαν και ποιες ενδέχεται να χαθούν που τις βλέπει αυτές τις θέσεις. Κύριε Να σας πω. Αυτό μας λένε για το πρόβλημα σε 11 διαφορετικές χώρες. Μεταξύ αυτών και η Βουλγαρία. Αλλά είναι και η Ρουμανία. Η χώρα του Επιτροπού Τσόλος. Ε, Ιταλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και η Φινλανδία. Όλες αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα που πλήττει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο διακυβεύεται εδώ είναι πάνω από 4.000 θέσει εργασία. Συν τα μέλη των οικογενειών τους που δεν θα έχουν μέσα να ζήσουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μεταρρύθμιση του 2006 είχε πράγματι σαν στόχο να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα των ζαχαρότευτων στην Ευρώπη. Και αυτή η μεταρρύθμιση έγινε με τίμημα σημαντικές θυσίε στο επίπεδο των ανθρώπων και των χωρών ή ε, περιφερειών. Ε, πολλές, πολλά εργοστάσια έκλεισαν και πολλέ περιοχέ εγκατέλειψαν την παραγωγή ζαχαρότευτλα η παραγωγή ε, ε, ε, ζαχαροκάλαμο, ζητούν την, μείωση, την κατάργηση όλων των δασμών. Ε, υπάρχει ένα προτιμησιακό καθεστώς προς τους παραδοσιακούς εταίρους μας. Η αγορά ζάχαρης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εντελώς ανοιχτή τα συμφέροντα των χωρών και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν ε, το αίτημα των ε, παραγωγών να τους ε, παρακάμψουμε. Η συνέλευσή μας έχει διαβολευτεί ε, πάρα πολλέ φορές, ειδικά σε σχέση με την έκθεση ΔΕΣ το 2011 και το ψήφισμα ε, του 2010 το οποίο ψηφίστηκε το 2011. Πράγματι χρειάζεται μια μεταρρύθμιση της απασχόλησης. Αλλά δεν θα πρέπει να επιταχύνουμε την ερήμωση της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Το Κοινοβούλιο εδώ και τρία χρόνια έχει επικυρώσει κατ' επανάληψη τη βούλησή του να προαπιστεί τα συμφέροντα των παραγωγών μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η αντιπρόσωπος Ρέντινγκ ε, δεν είναι η μόνη παρούσα εδώ που ε, δεν ξέρει πολλά πράγματα για την Γεωργία. Δεν είχαμε πραγματικά αποτελέσματα για τους παραδοσιακούς ε, παρασκευαστές ε, κατεργασμένης ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Ε, Δόθηκαν 5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008 στους παραγωγούς ζαχαρότευλους ε, σε σχέση με τους παραγωγούς ζαχαροκάλαμου είναι πολύ μικρότερο και αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν είναι ανταγωνιστικά. Έχει ε, υπάρξει μείωση της ε, προμήθειας ε, όχι γιατί ε, δεν ε, υπήρχαν ε, κατάλληλες δυνατότητες αλλά γιατί δεν επεκτάθηκαν όπως έπρεπε. Κάποιοι επιρρύπτουν ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. η μεταχείριση στους παραδοσιακούς ε, παραγωγούς ε, ζαχαροκάλαμου είναι άδικη και πραγματικά το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να είναι προκαταλημμένοι κατά όλων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα στον κατάλογο των ομιλητών, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Άλεφτσακ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, η πολιτική για τη ζάχαρη έχει αποτύχει πληρώνουμε περισσότερο για τη ζάχαρη από την παλιά. Σε ορισμένα μάλιστα κρατημέλη η βιομηχανία εξαφανίστηκε. Ξεριζώθηκε. Σε μερικές περιοχές παραδοσιακούς παραγωγούς ζαχαρότευτλου η οικονομία κατέρευσε. Η παραγωγή εξαφανίστηκε. Ήμασταν εξαγωγή και τώρα αγοράζουμε πάνω από 300.000 τόνους το χρόνο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδεύει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μας λέει απελευθέρωση η αγορά, εξού και το ερώτημά μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκτιμά ότι αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο τις δυνάμεις που κυριαρχούν στην αγορά και καταστρέφουμε τους μικρούς. Δεν θα ήταν καλύτερο να τροποποιήσουμε σταδιακά το παρόν σύστημα για να αποφύγουμε και τους κραδεσμού στην αγορά. Και τέλος, δεν θα ήταν καλύτερα να τροποποιήσουμε προοδευτικά τα όρια αυτά αντί να απελευθερώσουμε απότομα τον τομέα. Ευχαριστούμε. Θα έρθουμε στον κύριο... Θα περάσουμε στον κύριο Μάρζη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, στη συζήτηση αυτή για τη ζάχαρη θα ήθελα να ευθύσω την προσοχή σας στην ειδική κατάσταση των εξόχως περιφερειακών περιοχών που είναι σε δινή θέση μετά από την μεταρρύθμιση του 2005 και τώρα σε ακόμα χειρότερη θέση εάν δεν υπήρχαν οι αντισταθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Όπως γνωρίζετε, στα νησιά αυτά οι καλλιέργειες είναι ευάλωτες και πρέπει να προστατευτούν από τα καταστροφικά αποτελέσματα της επικείμενης, της επαπειλούμενης μεταρρύθμισης μετά το 2013 λόγω και των κανονών του ΠΟΕ. Γι' αυτό και καλό το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Γεωργίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν υπόψη τους την ειδική κατάσταση αυτών των ιδιαίτερως περιφερειακών περιοχών. Στην Ερεουνιόν είχαμε τρία εργοστάσια ζάχαρης και μένουν μόνο δύο πλέον. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νικολέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα του τομέα της ζάχαρης είναι πολύ ευρύτερο από τα όσα συζητούμε σήμερα και δεν ε, περιορίζεται μόνο στη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Η Ρουμανία, για παράδειγμα, έχει ε, αρκετή επάρκεια ζαχαροκάλαμου για την παραγωγή μόνο το 24% της ε, παραγωγής ε, που χρειάζεται και αυτό περιορίζεται από τις πεσοστώσεις και το υπόλοιπο ποσοστό διασφαλίζεται από την εισαγωγή ζάχαρης ακαταργαστής από το ζαχαροκάλαμο. Στο παρελθόν δεν υπήρχε πρόβλημα για την προμήθεια πρώτης ύλης ούτε και στη θέση της στην αγορά για τη Ρουμανία αλλά η ποσόστοση σημαίνει ότι έχουμε πολύ αυστηρά όρια για τις ε, πηγές πρώτων υλών ε, ακατέρδης ζάχαρης και δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ροή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει με κάποιο τρόπο τη μακροπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη επιβίωση των ε, παραγωγών ζάχαρης ε, και αυτό σημαίνει ότι ε, υπάρχουν εργοστάσια τα οποία ε, λειτουργούν στο πλήρες των δυνατοτήτων τους και παρόλα αυτά δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος τους δεν μπορεί να εισάγεται συνεχώς ακατέργαστη ζάχαρη. Θα πρέπει να ληφθούν κατεπίγοντα μέτρα ε, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διατηρήσει την εισαγωγή της, ε, ε, αλλιώς θα πρέπει να εισάγει όλη την ποσότητα ζάχαρης που έχει. Η ώρα είναι ιδιαίτερω προχωρημένη και θα ήθελα να δώσω το λόγο μόνο σε εκείνους που μέχρι στιγμής δεν συμμετείχαν στη συζήτηση. Είναι τρεις συνάδελφοι ε, ο κύριος Γιάρ πρώτος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά θα ήταν ε, το καλύτερο εάν δεν χρειαζόμαστε για τα ζαχαρότευτλα κανέναν κανονισμό αγοράς. Και βεβαίως ε, η κάθε ρύθμιση των ποσοστώσεων προσκρούει σε αντιστάσεις. Από την άλλη υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την ε, εξέλιξη των παγκόσμιων ε, τιμών. Γι' αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί μια ρύθμιση σχετικά ε, με ποσοστώσεις. Ε, θεωρώ ότι αυτή η απόφαση είναι σωστή. έχουμε το ζήτημα της παραγωγής από ισογλυκόζη, ε, ζάχαρης από ζαχαροκάλαμα και από ζαχαρότευτλα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των τριών αυτών μορφών παραγωγής, ώστε να υπάρξει κάποια σταθερότητα σε αυτό το τομέα. Βεβαίως θα ήταν ε, καλύτερα αν δεν χρειαζόμαστε το καθεστώς των ποσοστώσεων, αλλά νομίζω ότι προς όφελος των παραγωγών μας θα πρέπει να παρατείνουμε το καθεστώς των ποσοστώσεων. Σε ορισμένες ε, χώρες μέλη η ζάχαρη έχει γίνει ένα προϊόν ε, το οποίο σπανίζει γιατί και οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σε ύψος. Ε, αυτό δείχνει ότι ήταν αποτυχία η μεταρρύθμιση της αγοράς το 2006 και ε, στη δική μου χώρα έκλεισαν όλα τα εργοστάσια, χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τις θέσεις εργασίας τους και είναι σημαντικό να αλλάξουμε αυτή την ε, κατάσταση η οποία βασίζεται σε εσφαλμένες αποφάσεις του παρελθόντος και θα πρέπει να προσαρμόσουμε κάποιες ε, ε ρυθμίσεις, θα θυμίσουμε αυτή την κάμψη στον τομέα της ε, ζάχαρης. Η Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να ενισχύσει την απασχόληση και τη μεγέθυνση. Νομίζω θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις ισχύουσες διατάξεις για τις ποσοστώσεις. Ευχαριστώ κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης ε, που έγινε το 2006-2007 μας δείχνει τώρα πόσο περιορισμένη ήταν. Η αγορά, η παραγωγή ζάχαρης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μειωθεί σημαντικά και τώρα πολλές χώρες ε, χρειάζεται να εισάγουν ζάχαρη ενώ στα προηγούμενα χρόνια ήταν καθαρή εξαγωγής. Το ίδιο ισχύει και για τη Ρουμανία, διότι πλέον δεν μπορεί να καλύψει την εσωτερική τη ζήτηση με τα ε, χώρια ποσοστά παραγωγή. Η μελλοντική λοιπόν κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να λάβει υπόψη όλων αυτού του παράγοντε και θα πρέπει να προσαρμοζεί το σύστημα των ποσοστώσεων ώστε να δημιουργήσει παραγωγή και να έχουμε κατάλληλα επίπεδα ανάλογα με τη ζήτηση στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει επίση να εγγυηθούμε ε, θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων παραγωγής, ε, ε, παραγωγών ζάχαρης. Εδώ αναφέρομαι σε εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης ζαχαροκάλαμου που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα για την κατάλληλη προμήθεια. Υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Τη δέχεστε. Παρακαλώ κυρία συνάδελφε. Βρισκόμαστε ενώπιον μια τόσο σοβαρή κατάσταση, όπω αυτή που βιώνετε εσεί στη Ρουμανία ή όπω αυτή που βιώνουμε εμεί στην Πορτογαλία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να περιμένουμε να υπάρχουν μέτρα που θα επιτρέπουν παρέμβαση στον τομέα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική και να υπάρξει και μεταρρύθμιση στην κοινή οργάνωση αγορά ζάχαρη. Ε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, διότι θα χρειαζόμαστε και άμεσα μέτρα τα οποία θα μα επιτρέπουν να ε, φροντίσουμε τον τόπο. Κύριε Πρόεδρε, δεν είπα ότι δέχομαι το ερώτημα από τη συνάδελφο. Λυπούμε, αλλά είναι πολύ αργά και είμαι πολύ κουρασμένη. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην Επίτροπο την κυρία Ρέντινγκ για τις ε, τελικές της ε, παρατηρήσεις. Πρόεδρε, η συζήτηση κατέδειξε την διάσταση απόψεων μεταξύ των παραγωγών τεύτλων και από την άλλη μεριά των εργοστασίων ζάχαρης που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη εισαγόμενο ζαχαροκάλαμο. Οι πρώτοι μετά την μεταρρύθμιση προέβησαν σε μεταρρυθμίσεις, σε αναδιάρθρωση, με κόπο και κόστος, έγιναν όμως πιο ανταγωνιστικοί. Αυτοί που παραπονούνται σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι ακόμη δεν έχουν πάρει τις δύσκολες αποφάσεις. Είναι καιρό όμω να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Διότι αυτοί είναι οι κανόνες που συνομολογήσαμε. Η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μην έχετε καμία αμφιβολία. Η Κομισιόν θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τον ομαλό εφοδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς σε πρώτη ύλη. Το 2005 οι εισαγωγές ανήρχοντος σε 2,3 εκατομμύρια τόνους, σήμερα σε 2,5 και 3,1 εκατομμύρια τόνους. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ περατώνεται η συζήτηση. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο στις 12 Σεπτεμβρίου και θα ξεκινήσει στις 9. Ε, τα, η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί, ε, διατίθεται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και λύεται η συνεδρίαση. Καληνύχτα σας.